I um, have a number of announcements before we start. Um, I have received from the Council its position. Ανακοίνωση Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί στα πρακτικά ε, της συνεδρίασης. Η ε, τρίμηνη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κάνει γνωστή τη θέση στο Κοινοβούλιο αρχίζει από αύριο 21 Μαΐου 2010. Δεύτερον, τα χθεσινά ε, συνοπτικά